Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Έχουμε μία κάπως ε, ιδιόμορφη συνεδρίαση με ένα και μόνο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πέρα δηλαδή από την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Προέδρου, δεν έχει καφέ σήμερα. Και αυτό λόγω των απεριών δηλαδή. Και όχι λόγω μεθόδων λιτότητας. Παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία. Έχετε τον κατάλογο των γλωσσών εργασίας, χαιρετά τους διερμηνείς ο πρόεδρος. Ευχαριστούν οι διερμηνείς. Ο πρέπει να ετοιμάσετε και τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, εγώ ξέχασα τη δικιά μου στην Ολομέλεια βέβαια, για να μπορέσουμε να ψηφίζουμε τάχιστα. Θα υπάρξουν ψηφοφορίες που θα διασπάσουν την Επιτροπή μας. Χρειάζεται λοιπόν να προσφύγουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε εδώ για να ψηφίσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής Προϋπολογισμών για να προετοιμάσουμε δηλαδή την ψηφοφορία της επόμενης Ολομέλειας του Απριλίου 1 για τα προβλεπόμενα έσοδα και δαπάνες του Κοινοβουλίου για το 2012 έκθεση του κυρίου Φερνάντες. Είχαμε δύο συνεδριάσεις συνδιαλλαγής και προσυνδιαλλαγής με το Προεδρείο. Ε, βρέθη μία συμφωνία μεταξύ της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής του Προεδρείου υπό τους δύο αρμοδίους αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Αυτό έγινε πριν από δύο μέρες κατά τη δεύτερη συνεδρίαση διαβούλευσης την Τρίτη. Στη συνέχεια το χθεσινό Προεδρείο ενέκρινε τον προσωρινό προπολογισμό ενέκρινε τα προβλεπόμενα έσοδα και σήμερα και εμείς θα ψηφίσουμε γι' αυτά. Η ψηφοφορία στο Προεδρείο κάλυψε όλη την συμφωνία. Τις θέσεις που εμείς δηλαδή εκπροσωπήσαμε ως αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο εισηγητής προετοίμασε έναν συμβιβασμό που τροποποιεί την αρχική πρόταση συμπεριλαμβάνοντας τους όρους συμφωνίας. Ο εισηγητής φυσικά δεν θα συνενέσει σε εκείνες τις τροπολογίες που αντιβαίνουν τη συμφωνία αν είναι συμβατές οι τροπολογίες ο εισηγητής θα μας πει μάλιστα να τις ψηφίστε αν όχι θα πει όχι τώρα εμένα πρόθεσή μου όπως έχει υποδειχθεί δηλαδή και στον κατάλογο ψηφοφοριών να ψηφίσουμε καταρχήν τον συμβιβασμό αριθμό 1 που αφορά στην τρίτη παράγραφο, δηλαδή για την αρχή της συνολικής συμφωνίας υποστήριξη δηλαδή της Επιτροπής προϋπολογισμών προς τη συμφωνία εκείνη η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αντιπροσωπείας που την αντιπροσώπευσε παρά το Προεδρείο, αν απορριφθεί μετά θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά άμα περάσει τότε θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τις άλλες συμβιβαστικές προτάσεις και τις τροπολογίες. Κύριε Ισηγητά, θέλετε να μας πείτε πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για την συνεργασία τους και όλους ιδιαίτερους τους ε, σκεώδες εισηγητές γιατί στο στη σύντομη χρονική περίοδο Υπήρξαν διάφορες δυσκολίες ε, στη συνεργασία και στην επικοινωνία και γι' αυτό τους ευχαριστώ για την προσπάθεια που κατέβαλαν και φτάσαμε έτσι σε μια καλή συμφωνία συμφωνία στο Προεδρείο και στην Σε Ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις ε, τροπολογίες, για όλη τη συνεργασία και επίσης χάρη σε αυτή την παρέμβαση των πολιτικών ομάδων καταφέραμε και των ε, σχεδόν εισηγητών δηλαδή, καταφέραμε να φτάσουμε στο 2,3% αύξηση που στην πράξη είναι μείωση γιατί ο πληθωρισμός που χρησιμοποιεί η διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι στο 2,8%. Είναι προφανέ ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τώρα την συμφωνία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τις δαπάνες ούτε τις, ε, τα, τα έσοδα. Είναι θέμα συμβατότητας. Να κάνω μόνο μία διάκριση. Μπορεί να γίνουν εξοικονομήσεις μετά από τη συζήτηση. Εγώ ίδιος κάνω μια συμβαστική πρόταση έτσι ώστε σε ορισμένους ε, τομείς να γίνουν ε, εξοικονομήσεις. Αυτή η πρόταση είναι μια τροποποίηση της ALDE, ε, μια τροπολογία που είναι νομίζω η 17 όπου Αυτή η τροπολογία είναι συμβατή διότι πραγματικά αναζητά εξοικονομήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης. Έπειτα, οι σοσιαλιστές προτείνουν μια συμβιβαστική λύση. Στην προηγούμενη εκδοχή ήταν η υπαριθμόν 14 και τώρα είναι η συμβιβαστική υπαριθμόν 10 που, έχει, που αναφέρεται στην παράγραφο 14. Αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να το αποκαλέσουμε αυτό συμβαστική λύση, εγώ θα το πρότεινα καλύτερα ως προφορική τροπολογία. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα πρέπει να επιληθεί αυτό το θέμα γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά ε, και διορθώσεις στο αρχικό κείμενο και ήδη μπορούν να γίνουν και αφορούν το εκτιμώντας ε και επίσης στην παράγραφο 2 για να διορθωθεί το ποσό που είναι 1773 εκατομμύρια και 554.000 ευρώ. Αυτά τώρα είναι τεχνικές διορθώσεις. Θα μπορούσαν να γίνουν ήδη εξ αρχής, να μην είναι τροπολογίες και έτσι να έχει λυθεί αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Γκόραν Φέρμα ζήτησε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φινάνδε που προσπαθούμε να πετύχουμε έναν σφαιρικό συμβιβασμό εδώ. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε με τα αποτελέσματα τη ενδιαλλαγή. Για τεχνικού λόγου, νομίζω όμω ότι θα πρέπει το αποτέλεσμα τη συνδιαλλαγή με τα στοιχεία, τα αριθμητικά, θα πρέπει να είναι παραρτημένα στο κείμενο για να έχουμε κοντά μας τα αριθμικά σχέδια για να ξέρουμε ακριβώς τι δεχθήκαμε. Όπως είπε και ο κ. Φερνάντες, ακριβώς θεωρούμε ότι η πρότασή του για την συμβαστική τροπολογία 10 δεν είναι πραγματικός μια τροπολογία και γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Τέλος, το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί είναι ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπου υπάρχουν πολλά σημεία που δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη γνώμη στη συμβαστική πρόταση. Θα ήθελα να σας προτείνω, Πρόεδρε, λοιπόν, να ψηφίσουμε την δική του συμβαστική πρόταση, αλλά και τα συμπληρωματικά σημεία που θα θέλουμε να συμπεριληφθούν. Ιδίω για τη διαδικασία λήψη αποφάσει και για την γραμμή του προπολογισμού για τον οίκο αυτό τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ευχαριστώ, κύριο Μπόκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα μια που δεν είχα προσκληθεί στην συνάντηση με το Προεδρείο, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τους συμβασμούς. Ε, ευχαριστώ τον Πρόεδρο που θα ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες μία προς μία άσχετα από τις συμβαστικές τροπολογίες και επιμένω σε αυτό. Ευχαριστώ και ο Σαλβάρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που είπε ο κ. Σπόκος είναι λυπηρό και είναι πολύ λυπηρό ότι άμα από κοινού υποβάλλουμε τροπολογίες δεν μπορούμε από κοινού να διαπραγματευτούμε. Ελπίζω να γνωρίσει ο κύριος Βόκος ότι οι τρεις ομάδες με τις οποίες είχε συνυποβάλει κάποιες τροπολογίες δεν είναι υπεύθυνε γι' αυτό. Ε, βέβαια έχουμε μια κοινή ευθύνη γιατί ο στόχος μας είναι να πετύχουμε μια λύση. Ξέρω τους συνάδελφοι και της Γκου και των Πρασίνων στις συζητήσεις μας και για τους συμβασμούς ήταν παρόντε και μπόρεσαν και μάλιστα να ε, συμβαστούν. Θεωρώ ότι η πρόταση του κ. Μπόγκος αν τη δεχτεί ο πρόεδρος είναι λογική και θα έλεγα ε, όταν ε, ψηφίσουμε πάνω στις τροπολογίες να προσαρμοστούν τα αριθμητικά στοιχεία, οι αριθμοί δηλαδή των τροπολογίων μετά τις περικοπές που έγιναν. Γιατί όλες θα υπάρχει τελεία σύγχυση και δεν ξέρω από τεχνικής πλευράς τι λύση μπορεί να επιληθεί. Ευχαριστώ. Δεν θα τεθεί το πρόβλημα αγαπητέ φίλε. Θα ψηφίσουμε τους αριθμούς ε, στο παράρτημα. Ε, εκτός πια και αν ε, απορριφθεί ο συμβιβασμός, οπότε ξεκινάμε από την αρχή. Ο κύριος Πόρτας, ο οποίος έπαιξε το, το ρόλο του κακού στην ιστορία. Αυτό που είπατε ε, δεν ξέρω τώρα είναι αλήθεια κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα, το πρόβλημά μου είναι το εξής. Εκτός που δεν αναγνωρίζω του, οι συμβαστικές λύσεις που προτείνονται και άρα η ομάδα μου θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία, εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Συμβουλεύτηκα τον κανονισμό των Ευρωβουλευτών που στο 7ο άρθρο δίνει δικαίωμα σε διαβούλευση και σε ενημέρωση για όλους τους φακέλους, για όλους τους Ευρωβουλευτές και διαπίστωσα το εξή. ότι στο καταστατικό του βουλευτή δεν υπάρχει κανένα άρθρο ή παράγραφος σχετικά με την Τη μαριθμική αναπροσαρμογή οποιασδήποτε δαπάνης που έχει να κάνει με εμά με τον πληθωρισμό. Καμία δηλαδή τη μαριθμική προσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό σε σχέση με τις δικές μας δαπάνες. Με ένα άρθρο σε καμιά παράγραφο. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλες αυτές οι αποφάσεις για θέματα τη τη αναπροσαρμογής μισθή με επιδόματα ε, ε, ε, σπουδών, επιδόματα απόστασης, γενικές δαπάνες, όλα αυτές τα, οι δαπάνες ή τη μαριθμική τους αναπροσαρμογή απορρέει από αποφάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και το έγγραφο μέτρα εφαρμοστικά του καταστατικού που εγκρίθηκε στις 19 Μαΐου και στις 9 Ιουλίου του 2008 το οποίο τελευταία τροποποίηση είναι η 14η ε, Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Δηλαδή, όλα τα ποσά, τα κονδύλια που σχετίζονται με εμάς και επί των οποίων έχω κάνει μια σειρά από τροπολογίες που προτείνω μηδενική αύξηση για το 2012. Όλες αυτές οι τροπολογίες, χωρίς εξαίρεση, απορρέουν από αποφάσεις του Προεδρείου και δεν έχουν καμία σχέση με το καταστατικό του βουλευτή. Και γι' αυτό θα ήθελα να ειδοποιήσω όλους τους ε, συναδέλφους ότι όταν θα ψηφίσουν συμβιβαστικές ε, λύσεις που ως μόνο κανόνα έχουν να εξοικονομήσουν ε, από τα πάντα εκτός από αυτά που μας αντιστοιχούν εμάς να ψηφίσουν εν πλήρη γνώση της κατάστασης. Δηλαδή, θα υπερασπίσουμε τα δικά μας, ε, τα δικά μας έσοδα εναντίον των φορολογουμένων. Αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ για αυτή την επεξήγηση ψήφου και για αυτή την νομική επεξήγηση. Η Ελιζαμπέτ Ντουρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Έλγα Τρίπελ έχει καταθέσει ε, μια σειρά από τροπολογίες. Ε, συμφωνώ με τον ε, κύριο Άλβαρο. Τώρα η διαδικασία που μας προτείνεται σήμερα δεν μου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαφανής. Είναι δύσκολο να την παρακολουθήσουμε. Τώρα για την συνολική πολιτική εμείς θα σας ακολουθήσουμε. Τώρα αυτές τις τροπολογίες δεν τις υπογράψαμε για να μπορέσουν να περάσουν. Ωραία. Ευχαριστώ. Εκφράστηκαν όλοι οι συντονιστές εκτός από το ΠΠΕ αλλά κατανοώ ότι η σιωπή του ΕΛΚ σημαίνει την υποστήριξη προς τον εισηγητή. Ωραία. Προτείνω να πάρουμε την voting list. Τώρα, λόγω μου είπανε ότι επειδή είναι πολλοί οι παρόντες από το ΕΛ εγώ δεν έχω δικαίωμα ψήφου, άρα δεν θα ψηφίσω. Για τον ε, Προέδρε, συγγνώμη, Ξέχασα την κάρτα μου, έρχεται όπου να είναι. Αλλά μέχρι να έρθει η κάρτα μου, αν θέλετε να ψηφίσετε στη θέση μου. Αγαπητή Μπάρμπαρα, ούτε κι εγώ έχω την κάρτα μου. Λοιπόν, οπότε θα σας αφήσω να ψηφίσετε διανατάσεως της χειρός. Είμαστε οι δύο κακοί μαθητές αυτής της Επιτροπής, εγώ και εσείς. Συμβιβασμός 1, υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Πέντε. Σας ευχαριστώ. Αποχέ. Καμία. Αυτή η αίθουσα δεν είναι πολύ ευχάριστη ούτε για να οργανώνει κανεί συζήτηση ούτε να μετράει ψήφους αλλά η πλειοψηφία είναι σαφής. Λοιπόν, συμβιβασμός 2 για την παράγραφο 1 υπέρ κατά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αποχές καμία εγκρίνεται καταπίπτουν η τροπολογία 6 καταπίπτει Α, η 7 έχει αποσυρθεί. Ωραία, κάνε μας τώρα την τεχνική τροπολογία. Τεχνική τροπολογία. Για την παράγραφο 2. Είχα ζητήσει επίσης μια τεχνική τροπολογία για το εκτιμώντας ε. 16 Μαρτίου και 20 Μαρτίου να βάλουμε Τώρα για την παράγραφο 2 για τα νούμερα. Είναι 1773, 560, 543. Δηλαδή 1 δις 773, 560, 543. Πρόκειται για μία τεχνική τροπολογία επί του πρωτοτύπου για αυτές τις δύο τροπολογίες της τεχνικού χαρακτήρα όλοι συμφωνείτε φαντάζομαι κατά δύο αποχές εγκρίνονται ή οχτώ καταπίπτει διότι ήταν κατά της τεχνικής τροπολογίας τώρα συμβιβασμός 3 υπέρ Σηκώστε τα χέρια σας κατά. Τέσσερις κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται ο συμβιβασμός 3. Καταπίπτουν οι τρεις τροπολογίες 12 του κυρίου Βόγκαν. Είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Ένας. Δύο. Αποχές καμία. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Εκτός μικροφώνου. Α, η προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών για τον συμβιβασμό 4. Ο κύριος Πόρτας. Να προτείνω split vote, χωριστή ψηφοφορία. Διότι εγώ ήθελα να ψηφίσω κατά του πρώτου τμήματος. Για τον συμβιβασμό 4 λέμε. Και πού σταματάτε. Στην άνω Στην άνω το ελληνικό ερωτηματικό. Ο κύριος Φέρμε έχει μια προφορική τροπολογία. Ναι, θέλουμε να αφαιρέσουμε τη λέξη even. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε για το even, να διαγράψουμε το even. Κατά. Αποχές. Διαγράφουμε το even. Τώρα κατόπιν αιτήματος του κυρίου Πόρτας μέχρι την κοινοβουλευτική εφηβεία παραμένοντας κάτω από το πληθωρισμό. Je Ευχαριστώ. Κατά. Δύο κατά. Mm, très ε, ωραία, εποχές. Καμία εποχή. Το πρώτο εγκρίνεται λοιπόν. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο τη πρώτης. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχέ. Δύο αποχέ. Ε, λοιπόν. Το σύνολο, όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Adopted. Εγκρίνεται ο συμβιβασμός 4. Πάμε στην τροπολογία 17 του κυρίου Άλβαρο που είναι συμβατή αλλά δεν του αρέσει το εισηγητή. Να εξηγήσει. Ο κύριος Άλβαρο, πρώτο υπάρχει σύγχυση κύριε Πρόεδρε. Ε, και συνειδηθήκα με τον γιατί αυτή η τροπολογία δεν αφορά καμία άμεση περικοπή γιατί τότε θα έχουμε και προβλήματα συζητήσεις μας με τη γραμματεία του σώματος. Είναι κυρίως ένα θέμα εφαρμογής. Μόνο εφαρμογής. Δεν είναι περικοπή. Μόνο την εφαρμογή αφορά αυτό το σημείο. donc, le est pour. Είναι υπέρ τότε ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Ένας αποχές ουδεμία. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. 20 της κυρίας Ανδρεάσεν αλλά είναι κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Υπέρ. Δύο υπέρ. Κατά. Πολλοί άλλοι. Αποχές μία. Απορρίπτεται. 21 του κυρίου Βόγκαν και 22 είναι ακριβώς οι ίδιες. Και ο εισηγητής είναι κατά και των δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τσεκ. Ελέγχουμε. Δεν ψηφίζω εγώ και η Μπαρμπαρά θα ψηφίσει πώς αλήθεια. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, όλοι δεν ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ 18 κατά συγγνώμη ναι κυρία μου δεν δούλεψε το μηχάνημα τι ψηφίσατε υπέρ ή κατά κατά Λοιπόν, απορρίπτεται η τροπολογία. 19-18. Και οι δύο τροπολογίες, και 21 και 22, γιατί είναι ίδιες ακριβώς. Η 23 της κυρίας Ανδρεάσεν είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Τρεις. Κατά. Πολύ. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 του κυρίου Πόρτας είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Η αριστερά. Κατά. Ό,τι δεν είναι αριστερά. Αποχές πλειοψηφία κατά. 25 της κυρίας Βέρτμαν σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα να ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ εισηγητής υπέρ κατά ο κύριος Πόρτας αποχές καμία εγκρίνεται δεύτερο τμήμα δεν του αρέσει το εισηγητή υπέρ Τρεις. Κα, τέσσερις. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 28 Άλβαρο. Η συγκεκριτής είναι υπέρ. Alors, euh, monsieur rapporteur. Κύριε Σιγητά, θέλετε τον λόγο. Να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει αλλαγή και ότι όσον αφορά την εκτέλεση είμαι υπέρ. διότι διαφορετικά καταπίπτει. Donc, ça doit être Άρα λοιπόν θα πρέπει να ερμηνευθεί ω σχετικό με την εκτέλεση. Με αυτή την ερμηνεία ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Σα ευχαριστώ. Κατά. Οι σοσιαλιστέ. Μα είναι μόνοι του. Αποχέ. Δεν υπάρχουν αποχές, άρα εγκρίνεται. 29 καταπίπτει. Συμβιβαστική υπαριθμών 7. Ποιοι είναι υπέρ. Nous Τι θέλετε να το ψηφίσουμε. Όχι, μόλις το εγκρίναμε. Η 29 καταπίπτει, συμβαστική 7, υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά 5 abstention αποχές εγκρίνεται. Euh, Ce qui nous amène à l'amendement 41 de Madame. Και έτσι φτάνουμε στην τροπολογία 41 της κυρίας Ανδρέασεν. Ο εισηγητής είναι κατά. Όχι. Δεν κατάλαβα καλά. Στο 40. Στο 40 και εδώ πρέπει να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Ο εισηγητής πιστεύω πως το δεύτερο τμήμα της χωριστής ψηφοφορίας καταπίπτει. La deuxième partie... Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Και τι λέει το δεύτερο τμήμα? Το πρώτο τμήμα σταματάει εκεί που λέει οι υπηρεσίε της, ε, της ε, βιβλιοθήκης προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη στις τρεις γλώσσες εργασίας και το δεύτερο τμήμα καταπίπτει με βάση τις προηγούμενες ε, τροπολογίες που ψηφίσαμε δεν είναι συμβατή με τη συμβαστική λύση. Μάλιστα. Για το πρώτο τμήμα ο είναι ούτως ή άλλως κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν για το πρώτο τμήμα τη 40. Ποιοι είναι υπέρ. Je vous remercie. 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre Kata. Αποχές. Καταπίπτει, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει, δεν μένει τίποτα πλέον από την τροπολογία 40. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία 41. Ο κύριος Σαλβαρό έχει απελπιστεί. Εντάξει, μην στεναχωριέστε, θα κερδίσετε αλλε 41 Αντρέασεν. Ο εισηγητή είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Σας ευχαριστώ, αποχές, απορρίπτεται. 42 και 43 έχουν εξαφανιστεί και ψηφίζουμε για την... Όχι, ο κύριος Φέρμ. Δεν έχω πρόβλημα για την 42. Εγώ νομίζω πως πρέπει να ψηφίσουμε τις 42. Απλώς θέλω να εξηγήσω ότι η ομάδα μου θα καταψηφίσει παρά το γεγονός ότι συμπαθεί κάπως την 47 και την 50 και αυτήν εδώ γιατί είναι εσωτερικά αντιφατικές, γιατί ορισμένες από τις εσωτερικές δαπάνες λένε ότι θα πρέπει να είναι business class αν καταξιδεύει κανείς πάνω από 4 ώρες, ενώ άλλη, σε άλλη μεριά λέει ότι μόνο αν καταξιδεύει κανείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε το κόστος και τις δαπάνες των Ευρωβουλευτών, αλλά πιο οργανωμένα και πριν από τη δημοσιονομική διαδικασία του φθινοπόρου. Θα το καταψηφίσουμε τώρα δηλαδή, αλλά θέλουμε να ξαπανέλθουμε στο ζήτημα. Ευχαριστώ για τα οδηπορία Χρειάστηκε εγώ προσωπικά να κάνω μια πρόταση στη συνδιαλλαγή που δεν λήφθη όμω σοβαρά ούτε από τη δική μου αντιπροσωπή ούτε από αυτή του Προεδρείου αλλά μπορούμε να την ξαναδουλέψουμε για το φθινόπωρο. Ψηφίζουμε λοιπόν για τη 42 κύριε Μποκρός. Για τη 42. Όπως σα υποσχέθηκα. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. 6, 7, 8, 9. Qui est contre Un Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 43 όμως καταπίπτει. 44 Άλβαρο και λυπή και μπουκρός. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές, δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται. Η 45 έχει καταπέσει, 46 Ανδρέασεν, ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Πριν ψηφίσουμε, ε, ο εισηγητής θέλει το λόγο. Για το συμβασμό υπαριθμών 9, Πρόεδρε, έχω να πω ότι ζητώ και αυτό σύμφωνα και με την πρόταση του Πρόεδρου μας κατά την εκτέλεση να καταβληθούν προσπάθειες για να υπάρξουν μειώσεις στη χρήση ύδατος, ηλεκτρονισμού, χαρτιού, αλλά και για το κόστος μεταφοράς στις επίσημες αποστολές και το ταξίδι των βουλευτών. Αυτό είναι ο συμβασμός που προτείνω. Πρόεδρος, ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό λέει και το γραπτό κείμενο. Αυτή είναι μια επεξήγηση του περιεχομένου του συμβαστικού ε, κειμένου. Δεν είναι προφορική. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής εννέα. Ευχαριστώ. Κατά. εποχές. Εγκρίνεται. Σαραντοκτώ. Μποκρός. Ο ζήτης είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Ο κ. Άλβαρο έχει κάτι να πει. Ενδεχομένως για να είμαστε σύμφωνοι με αυτό που είπε ο κ. Μπόκρος εισαγωγικά και ταυτόχρονα να μην διακυβεύσουμε τους προθέσεις της ε, έκθεσης. Έχω να ρωτήσω αυτούς τους συναδέλφους που έχουν συνυπογράψει την τροπολογία. Θα συμφωνούσαν να αφαιρεθεί αναφορά στο 2011 γιατί αυτό αναφέρεται σε συμφωνία με το Προεδρία που προβλέπονται κάποιες περικοπές. Θα μπορούσαμε έτσι και στο μέλλον όσο αφορά το κόστος καθαρισμού ή διαχείρισης να συνεχίζουμε να προσπαθούμε να το μειώσουμε. Εάν βγάλουμε λοιπόν αυτή την αναφορά στο 2001 και συμφωνήσουν οι δύο συνυπογράφοντες, αυτό δεν θα είναι αντίθετο με τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε εκεί. Ταυτόχρονα μας θα λέμε συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μειώσουμε αυτό το κόστος. Δεν ξέρω τώρα η εισηγητής τι έχει να πάνω σε αυτό. Αλλά δεν θα ήταν αντίθετο με το συμβασμό, θα συνέβαλε όμως με αλληλεγγύη για να λύσουμε το πρόβλημα. Πρόεδρος. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε, αντί να πούμε, ε, επιτρέποντας να διατηρηθεί το επίπεδο δαπανών του 2011, εάν δεν έχει καμία αλλαγή να προσθέσουμε. Ο εισηγητής. Ο 48 καταπίπτει. Λόγω του συμβιβασμού. Αλλά για να επανέλθουμε θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε. Πρώτος, η προφορική τροπολογία του κυρίου Άλβαρο. Ναι, αρκεί. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι, παραμένει συνεπές το κείμενο. Ρωτάω λοιπόν τους δύο συνυπογράψατε, Δεχόσαστε την προφορική τροπολογία του κ. Άλβαρο, όπου θα ψηφίσουμε. Ο εισηγητής όμως μας είπε ότι είναι κατά ή όχι. Εγώ δεν έχω καμία επιλογή παρά να παραμείνω στην αρχική πρόταση και δεν καταλαβαίνω οι φιλελεύθεροι γιατί υποστηρίζουν τη δική του πρόταση. Μα προσπαθούμε να σα βοηθήσουμε, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, υποβάλλουμε την τροπολογία αυτή όσα έχει διατυπωθεί. Ο εισηγητή είναι κατά διότι δεν είναι συμβατή με την συμβαστική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ τη 48. Ο κ. Υποκρός είναι υπέρ. Μπράβο. Τρει. Τέσσερις. Ποιος είναι κατά. Κατά. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Άλβαρο αποχή. Με όρους ελεύθερος. Ωραία. Ωραία. Μπορούμε να δώσουμε 49. Τροπολογία Γκρέσλε. Ο εισηγητές είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Η Ψηφοφορία λοιπόν υπέρ της Ίνια. 50. Καταπίπτει όμως. Ο κύριος Πόρτας. Μα μια που πλη... ψηφίσαμε την 47 και υπάρχουν δύο μέθοδοι για να φτάσουμε τον ίδιο στόχο να ψηφίσουμε και την 50. Αν δεν διαφωνεί ο εισηγητής να ψηφίσουμε πάνω στις 50. Μα μου φαίνεται πρόεδρε ότι έχει καλυφθεί από τη συμβαστική τροπολογία που υπερψηφίσαμε που λέει ότι θέλουμε μείωση των δαπανών στις αποστολές. Ο κ. Σπόρτας. αυτή η συμβαστική είναι γενική φύση. Αυτό που προτείνει αυτή η παράγραφο είναι η συγκεκριμενοποίηση. Αφού ψηφίσαμε λοιπόν για την παράγραφο 47, είναι θέμα, 47 <coughs> είναι θέμα συνοχής. Πρέπει να ψηφίσουμε και αυτήν την μεταβλητή, που είναι απλώς πιο συγκεκριμένα το ίδιο πράγμα. Ωραία. Ψηφίζουμε για την 50. Ποιοι είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική δέκα λέει ο κατάλογος της που δεν είναι όμως πραγματική συμβαστική τροπολογία αλλά μια προφορική τροπολογία του εισιτή ποιος είναι υπέρ το ίδιο κείμενο είναι κατά Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Το κείμενο που αποκαλείται συμβαστική τροπολογία 10 ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Γιατί είναι μυστική ψηφορία. Ωραία, είναι μυστική, αλλά θα σας πω το αποτέλεσμα. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Ωραία. Πέρα ψηφορίας. 22 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Η 51 καταπίπτει λοιπόν. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Για να ξαναλέξουμε ηλεκτρονικά. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 17, 19 κατά, συγγνώμη. Εγκρίνεται λοιπόν. Κατά αυτό τροπολογίας μέχρι το 59 του κυρίου Φέρμ. Πρόεδρε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η αγαπημένη της τροπολογίας μας είναι συμβατό με την τροπολογία που εγκρίζαμε τώρα. Γιατί όσον αφορά σε μια πρότυπη διαδικασία του Κοινοβουλίου, διαφανή διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό να το ψηφίσουμε νομίζω ως προσθήκη. Έχω και μια προφορική τροπολογία που θα ήθελα να ψηφίσουμε. Που λέμε δεν, υποσ... δεν υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενό νέου συγκεκριμένου κονδυλίου για το οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Και να μεταφέρουμε το 1 που προβλέπτε στο 2007. Το σωστό θα ήταν όμως να πούμε όχι στο 2007 στο αποθεματικό. Θεωρεί όμως ότι οποιοδήποτε δημιουργία μιας τέτοιας ε, δημοσιονομικής γραμμής θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τις ε, επί του προπληκτισμού αρμόδιες αρχές. θα μας πει ο εισηγητής τι θέλει. Κύριε Σάλβερο, ήσασταν πάρα πολύ σίγουρα, ε, γρήγορος όλων. Λυπάμαι τους Ιερεμίες και ούτε και εγώ κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή τι θέλετε, να τις ψηφίσουμε μαζί την τροπολογία, να ενώσουμε ξεχωριστά. Κοιτάξτε, μα τις έχετε γραπτά. Και γι' αυτό ήμουν τόσο γρήγορο. Επαναλαμβάνω. Το, πρώτο λέει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη κοινοβουλευτική διαδικασία για την λήψη απόψη και ανοιχτή συζήτηση. Και γιατί, γιατί δεν θεωρούμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνουμε κάτι το διαφορετικό. Παρά μόνο να έχουμε την προπαρασκευαστική εργασία. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει στο τελικό πράσινο φως. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να εγκρίνουμε κάποια στιγμή αργότερα μία ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή. Αλλά όχι τώρα, γιατί αυτό δεν θα δίνουμε το πράσινο φως. Να το αναβάλουμε μέχρι τη δημοσιονομική διαδικασία το φθινόπωρο για να έχουν προχωρήσει τα πράγματα και να μπορούμε να αποφάσουμε. αποφασίσουμε. Συγγνώμη. Αυτό διαφανή μόνιμη διαδικασία και η γραμμή του προπολογισμού οριστεί όχι τώρα, μέσα στα πλαίσια τη δημοσιονομική διαδικασία του φθινόπωρο. Ωραία, λέει ο Θα δώσω το λόγο στον ζητητή. Προηγουμένως, όπω για να προσθέσω τα πράγματα, έχω να πω ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστέ τροπολογίε. Η μία είναι η 52, που υποβάλλει ο Γκέραν Φέρμ για να συμπληρωθεί Συμβαστική 11. Προσθήκη, έτσι. Λοιπόν. Και η δεύτερη πρόταση για τη δημοσιονομική γραμμή είναι η τροπολογία 59. Που θα ήταν επίσης προσθήκη. Εντάξει. Λοιπόν. Ο συγητής. Θεωρώ ότι όταν ψηφίσαμε το συμβιβασμό ο οποίος συνεκρίθη η τροπολογία 52 καταπίπτει. Και αν καταπέσει, δεν τίθεται θέμα και για μια νέα κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Άποψη είναι όμως ότι καταπίπτει. Γιατί μία συμβαστική τροπολογία οδηγεί τις άλλες τροπολογίες για το ίδιο θέμα στο να καταπέσουν. Για την παράγραφο 15α, τροπολογία 59, ε, θα υπάρξει μια προφορική τροπολογία. Για να μην είμαστε αντίθετοι στη σφαιρική συμβαστική τροπολογία που υιοθετήσαμε. Αυτό κατά γνώμη μου. Το πρώτο δηλαδή που πρέπει να εξετάσουμε είναι κατά πόσον καταπίπτει 52 ή όχι. Νομίζω ναι. Και υπήρχε στο κατάλογο της ψηφοφορίας και κανένας από τις πολιτικές ομάδες που γνωμοδότησαν για άλλα σημεία δεν είπαν τίποτα μέχρι στιγμής σχετικά με το αν υιοθετηθεί η 11, η συμβαστική 11, άλλε τροπολογίες δεν θα καταπέσουν, ενώ αναφέρεται αυτό το κατάλογο ψηφοφορία. Πρώτος, η Μόνικα Χολμάιερ και μετά ο Γκέραν Φέν, η Μόνικα. Επί της ουσίας, Πρόεδρε, θέλω να πω στον Γκραμ Φέρμ ότι θα υπάρξει μία κοινοποίηση. Αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία. Δεν αποφασίσαμε ποτέ ότι θα κάνουμε μία, θα ακολουθήσουμε μία κανονική διαδικασία, αλλά θα το κάνουμε. Αν δεν υπάρχει κοινοποίηση δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τον Ευρωπαϊκή Ιστορία, γιατί θα ήταν παράνομο. Και έχει συμφωνηθεί αυτό. Μία συνήθεια διαδικασία που θα μας απασχολήσουν εδώ. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, θα υπάρξει αυτή η διαδικασία κοινοποίηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το ψηφίσουμε. Θα γίνει αυτό, γιατί είναι υποχρεωτικό από νομικής πλευράς. Και μετά μπορούμε να το σκεφτούμε μέσα στα πλαίσια της συμφωνώ να υπάρχει μια ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό γιατί νομίζω ότι αυτό αυξάνει την διαφάνεια, δεν τη μειώνει. Εγώ πάντως αφορά τα μεγάλα σχέδια ήθελα μια ξεχωριστή γραμμή στον προπονισμό, γιατί έτσι ξέρουμε τι θα πανίσαμε και τι δεν θα πανίσαμε. Είναι λοιπόν υπέρ της αρχής της διαφάνειας. Και δεν ξέρω γιατί να μην θέλουμε να υπάρξει μια γραμμή στον προπολογισμό. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την κοινοποίηση. Je Εγώ νομίζω πως το εξήγησε αυτό πολύ καλά και στη τελευταία συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή. Καταρχήν πιστεύω πως αυτό εδώ δεν είναι μια κανονική διαδικασία λήψη αποφάσεων, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μόνο ένα κτηριακό πρόγραμμα, είναι κάτι παραπάνω και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι αρκεί αυτό που λέει η Μόνικα Χολμάγερ. Υπάρχουν και πολλές άλλες πτυχές εδώ που δεν το καταστούν ένα απλό πρόγραμμα ε, ε, ε, κτηριακό. Θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία που είτε θα έρθει κατευθείαν στην Ολομέλεια ή τουλάχιστον θα είναι τμήμα της κανονικής δημοσιονομικής διαδικασίας που εγκρίνεται από την Δημοσιονομική Αρχή που θα το κάνει το φθινόπωρο και όχι στις εκτιμήσεις. χωριστή γραμμή. Δεν είμαι κατά. Είμαι υπέρ. Αλλά όχι στις εκτιμήσεις. Θέλω να είναι αυτό το τμήμα τη φυσιολογική δημοσιονομική διαδικασία που εγκρίνεται από τη δημοσιονομική αρχή και να είναι απόλυτα διαφανέ. Δεν είμαι κατά τη δημιουργία χωριστή δημοσιονομική γραμμή, αλλά όχι τώρα. Γιατί αυτή δεν είναι η κανονική διαδικασία για να φτιάχνουμε τέτοιου είδου γραμμέ. Και έχω πει στον εισηγητή αρκετέ φορέ ότι τα θέλω αυτά εγώ μέσα στην συμβαστική λύση και γι' αυτό δεν το δέχτηκε και γι' αυτό θέλω να τα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Όπως... Δεν ξέρω πώς λέγεται στα πορτογαλικά ή στα γαλλικά, αλλά συμβιβασμό στα γαλλικά θα πει ότι όλοι συμφωνούν. Και μας έρχονται εδώ τώρα τροπολογίες οι οποίες δεν είναι μέσα στο συμβιβασμό 11. Και μπορούμε κάλλιστα εμείς να επιχειρηματολογούμε και να λέμε ότι ναι, πρόκειται για ένα συμβιβασμό ο οποίος ασχολείται με τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας κλπ. <coughs> Αυτό όμως δεν μπαίνει μέσα. Από τυπικής απόψεως, το να λέμε ότι ήδη έχουν λυθεί, δεν είναι σωστό. Διότι πολιτικά υπόθηκε ότι το περιεχόμενο δεν συμπεριλαμβάνεται στην τροπολογία. Οι τροπολογίες 52 και 53 πρέπει λοιπόν να ψηφιστούν γιατί δεν καλύπτονται από το συμβιβασμό. Εγώ θέλω να υποστηρίξω το αίτημα των σοσιαλιστών διότι πέρα από την ε, μορφή γι' αυτό το σχέδιο το οποίο εγώ είμαι μια, το οποίο εγώ είμαι μια μεγάλη οπαδός πιστεύω ότι θα πρέπει να συσπηρωθούμε και να τα βρούμε όλοι γύρω από αυτό το σχέδιο Πρέπει λοιπόν όλες οι ευαισθησίες, όχι μόνο οι δημοσιονομικές, αλλά και αυτό το οποίο βάζουμε πίσω από το δημοσιονομικό, πρέπει να συσπηρωθούν για να προχωρήσουμε στην όσο το δυνατόν σωστότερη και καλύτερη οικοδόμηση αυτού του σχεδίου στους επόμενους μήνες. Ωραία, προτείνω να ψηφίσουμε την τροπολογία 52 πρώτα ως συμπλήρωμα. Δεν ψηφίζω γιατί δεν έχω το δικαίωμα, έχει πολλούς πεπέ. Προτείνω στους συντάκτες της τροπολογίας μία προφορική τροπολογία αναφέρεται ότι όλες οι αποφάσεις που συνδέονται με το σχέδιο πρέπει να υπόκεινται στην πάγια κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι στην appropriated, στην κατάλληλη, στη σωστή. Εμείς λέμε standard, δηλαδή στην πάγια κοινοβουλευτική διαδικασία. Συμφωνείτε, ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 52 με τη λέξη από το standard αντικαθιστούμε το appropriate. Είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ. Κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία κατευθείαν. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται η τροπολογία. Οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν μέχρι την 59 και εκεί έχουμε πάλι την 59. Η 59 για τη γραμμή του προϋπολογισμού. Είναι κατά ο εισηγητής κατευθείαν. Α, ο εισηγητής έχει το λόγο. Νομίζω ότι... επειδή υπάρχει ένα συμβιβασμός, αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε ένα συμβιβασμό μπορούμε να, να χώσουμε τη θέληση του καθένα και τις επιθυμίες του. Θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε σε αυτή την παράγραφο και να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ένα σχετικό άνοιγμα οριζόντων για να έχουμε μια μεγαλύτερη συνένεση. Τι θέλει να πει αυτό κύριε Σιγητά, αλήθεια. Λοιπόν, Προτείνω να ψηφίσουμε καταρχήν την 59. Είναι υπέρ ή κατά ο εισηγητής. Κατά. Ή ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τροπολογία 59. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ 15 κατά, άρα περνάει η 59. Λοιπόν, να θεωρήσουμε κύριε εισηγητά ότι λόγω αυτών των αντιφατικών ψηφοφοριών, άρα πολιτικά συμπληρωματικών, ε, το πολιτικό πνεύμα προσεγγίστηκε Τροπολογία 1 της κυρίας ενώ ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Ευχαριστώ, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 της κυρίας Βέρτμαν είναι υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλιστές. Αποχές πλειοψηφία υπέρ. τρία συμβατή με τη δύο αλλά είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Υπέρ της τρία Κατά. Απορρίπτεται. τέσσερα είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τεχνική τροπολογία του εισηγητή που ήδη την ψηφίσαμε και οι πέντε της κυρίας Ανδρεάσαν υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Δεν ψηφίζω εγώ. Αλλά αρχίζει η ψηφοφορία και είναι μυστική. Πέρα στις ψηφοφορίες. 33 υπέρ κατά συγχαίρω τον εισηγητή ευχαριστώ τους συντονιστές και όλους όσους ετοίμασαν τους συμβιβασμούς πριν τελειώνουμε τη συνεδρίαση σιωπή τελείωσε η ψηφοφορία και όσοι θέλουν να πήγουν να πήγουν. αλλά δεν τελείωσε η συνεδρίαση γιατί στα any other business στα διάφορα η Ίγκε Γκρέσλε θέλει να κάνει μία ανακοίνωση και θα την ακούσουμε ήσυχα. Πρόκειται για το προεπολογισμό. Τη μέθοδο του προεπολογισμού θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα, γιατί η Κομισιόν έχει στείλει διάφορα non-paper στι ομάδε εργασία και φοβούμαι ότι υπάρχει πλήρη σύγχυση. Αυτά τα νόνε ε, ε, papers αφορά τις πράξεις, τις τιμές, τις υποχρεώσεις εκείνων που έχουν, στους οποίους έχει να τηθεί ε, η ευθύνη κλπ. Οι προτάσεις της Κομισιόν να αναπορίζει τα χρηματοδοτικά μέσα, το πλαίσιο, το ότι πρέπει να υπάρχουν κοινά συμφέροντα κλπ. Αυτά τα έχουμε εντάξει όλα. Στις εν πράξεις, τι έχει το θέμα κατά πόσον η εξοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί στην Κομισιόν και πώς θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην υιοθέτηση αυτών των κατεξιώσεων πράξεων. Η Κομισιόν μας έστειλε μία λίστα 117 σημείων 117 άρθρων για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει κατοξιδότηση πράξη. Εμείς ε, δεν ακολουθούμε 10 από αυτές απο 107 υπόλοιπες τις δεχόμαστε. Από την άλλη μεριά η Κομισιόν υπέβαλε τώρα και έγγραφα όπου λέει ότι θα πρέπει από το εκτελεστικό τμήμα να περάσουμε στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και εδώ θα την ακολουθήσουμε εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Τα άλλα όσον αφορά τα δικαιώματα της εξοδότησης δεν θα ακολουθήσουμε την ε, Κομισιόν και δεν θέλουμε να περάσει αυτό από τον δημοσιονομικό κανονισμό στο εκτελεστικό τμήμα. Αυτό ήθελα να το πω απλώς. Γιατί αλλιώς ε, τρομάζουμε όλοι τι να κάνουμε όλα αυτά τα έγγραφα. Λοιπόν, τα έγγραφα έχουν όλα ληφθεί υπόψη από την εισηγήτρια. Ήθελα να σα το πω απλώ προ την ενημέρωσή Σα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, εγώ σας ευχαριστώ. Άλλε ε, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Ευχαριστώ πέρα συνεδρίασης.